Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής των Προϋπολογισμών παρακαλώντας σας να μας συγχωρήσετε για την καθυστέρηση που οφείλεται στην ε, παράταση των εργασιών της συνεδρίας των συντονιστών λόγω βεβαρημένης μερισίας διτάξεως. Η ημερήσια διάταξη ελπίζω να εγκρίνεται. με την υποσημείωση ότι το σημείο 9 αναβάλλεται. Επαόριστο. Και το 14 για τη Frontex. Γιατί δεν λάβαμε τα έγγραφα που απαιτούνται για να λάβουμε θέση και βέβαια για τον εισηγητή μας Ραμουλμέιρ να διατυπώσει την πρότασή του. Αν δεν έχετε αντιρρήσει λοιπόν, και με την αναβολή αυτών των δύο θεμάτων εγκρίνεται η Μαρίσια διάταξη. Οφείλω να σας ενημερώσω για μια απόφαση που μόλις έλαβαν οι συντονιστές. Θα ζητηθεί άδεια για έκθεση πρωτοβουλίας σχετική με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχετε λάβει τα σχέδια πρακτικών. των ε, ημέρων των συνεδριάσεων 9η και 10η Νοεμβρίου, 9η Δεκεμβρίου, 9η και 12η Ιανουαρίου και 1 η Φεβρουαρίου. Αν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν, εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά και δίνουμε το λόγο στο συνάδελφο Ρίτσαρτ Ashworth, εισηγητή των λοιπόν τμήματων του σχεδίου προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έτος 2018. Σας ευχαριστούμε για το σχέδιο κύριε Σιγητά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης που έχετε μπροστά σας είναι το τρίτο σε αυτή την θητεία και στο πλαίσιο αυτού του ΠΔΠ. Και θα ήθελα εδώ πέρα να επενέσω τους δύο προκατόχους μου, τους κυρίους ε, Τάραντ και Ντεπρέ για την δουλειά που έχουν κάνει. Είχαν στείλει την προηγούμενη έκθεση στους και οδησηγητές και έχουν σωματώσει ήδη κάποιες παρατηρήσεις τους, αλλά τώρα δεν θα τα ξαναπώ όλα αυτά για λόγους συντομίας. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να αναφέρω τις προτεραιότητες ε, που έχω. Πρώτα απ' όλα, όπως πάντα, έχουμε ακριβώ ε, τον στόχο να διατηρηθεί ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου κάτω από το 20% του τίτλου 5 και για να γίνει αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε εξοικονομήσεις ε, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Προεδρείου. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους προτάσεις. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να επιτελέσει τις ε, λειτουργίες του και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό και τις ε, υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Αλλά τρίτη προτεραιότητα είναι το θέμα της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Σαφώς έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των Ιδρυμάτων. Θα ξέρουν οι συνάδελφοι πως έχουμε κάποιες πολύ γνωστές ε, περιπτώσεις ε, που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και έχουν αναδείξει κάποιες ε, αδυναμίες. Αυτό δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι επικρινώ όλα τα κόμματα και τα ιδρύματα. Μακράν αυτό. Εκεί όπου υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, ευχαριστώ να συνεχίσουν, αλλά Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία και άρα έχω εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό και εδώ πέρα οφείλω να επενέσω την διοίκηση για τα σχετικά μέτρα και πραγματικά πρέπει να τους στηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ε, τα άλλα ζητήματα τα οποία έχω αναφέρει πέρα από την ε, ασφάλεια πράγματι υπάρχει το ζήτημα των κυβερνοεπιθέσεων και βεβαίως εγώ εξακολουθώ να στηρίζω το θέμα της κυβερνοασφάλειας το τωρινό πολιτικό κλίμα είναι μια αυξανόμενη απειλή και πρέπει να έχουμε κατά νου τους κινδύνους ε, και καλό είναι να προτρέχουμε παρά να αντιδρούμε. Για τα κτίρια. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι απογοητεύτηκα για το ότι το Προεδρείο δεν χάραξε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που είναι παραδοσιακά μια δέσμευση την οποία αναλαμβάνουν αλλά τελικά δεν εκπληρώνουν. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουν σε μια τέτοια πρακτική και όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα για το κτίριο Adenauer και την κατασκευή του. Ε, είμαι υπέρα αλλά πρέπει να εξοδευτούν σωστά τα χρήματα για το κτίριο PHS και πάλι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, προτάσεις ε, του Προεδρείου Δεν τη ζήτημα ότι υπάρχει ένα θέμα με το κτίριο και Κάποια από αυτά τα λεφτά βεβαίως θα πάνε σε κάποιες προεργασίες, αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Μια που αναζητούμε λοιπόν εξοικονόμηση εντός του προπολίσμου του Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει είναι οι προφορικές επεξηγήσεις ψήφου. Δεν έχω πρόβλημα με το να κάνουν κάτι τέτοιο οι βουλευτές, αλλά αναρωτιέμαι γιατί εάν ε, αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση γιατί πρέπει να μεταφράζεται σε 23 διαφορετικές γλώσσες. Ε, Βεβαίω, γιατί όταν κάνουμε κάτι τέτοιο κάνουν άλλη μία βάρδια οι ομάδες των διερμηνέων, κάτι το οποίο κοστίζει. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή ε, στην οποία ενθαρρύναμε απλά τους βουλευτές και τους ε, δίναμε την δυνατότητα του Voxbox. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις μεθόδους ε, ή κάποια άλλη μέθοδο για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τέλος, για το πρόγραμμα επικοινωνίας για τις ευρωεκλογέ του 2019, ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε ε, χρήματα για να στηριχθεί αυτό το πρόγραμμα, το δέχομαι. Συμφωνώ ότι πρέπει να αρχίσουμε από τώρα τον προγραμματισμό και θα ε, ενθαρρύνω τους συναδέλφους να κοιτάξουν προσεκτικά το θέμα της κατανομής της δαπάνης αυτής και να παρακαλέσω τους συναδέλφους να προσπαθήσουν να βρουν πού, πώς και πότε θα ξοδευτούν αυτά τα λεφτά. Κάτι παρομοιό για το γενικό επίδομα των βουλευτών το επίδομα γενικών δαπανών. Είχα διάφορα αιτήματα για περισσότερη διαφάνεια, τα οποία ευχαρίστω θα στήριξω. Κύριε Πρόεδρε, θα συναντήσω και την πέμπτη τους σκιοδησίτες, αλλά αναμένω τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Ευχαριστώ. Κύριε θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Κάποιοι ήδη έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Ρουμπίχ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο. Βλέπουμε ότι ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα θέμα πολύ λεπτό. Ο Ρίτσαρτ νομίζω με τις παρατηρήσεις του το επισημαίνει πολύ εύστοχα. Εμένα με ενδιαφέρουν ζητήματα αρχής για την ενίσχυση της δημοκρατίας της Ευρώπης στο μέλλον. Με αυτό το 4% λιγότερο για τα επόμενα 7 χρόνια που μας έχουν επιβάλει οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων, έχουμε πρόβλημα, πρέπει να μειωθεί και κατά 1% επιπλέον το προσωπικό και βεβαίως για το 2018 με τις διαπραγματεύσεις του Brexit θα πρέπει να καλύψουμε επιπλέον εργασίες και λειτουργίες με περιορισμένο προπολογισμό, χωρίς να ξέρουμε τι είδους λύση, εάν μπορέσει να βρει, θα δώσει η πολιτική ηγεσία. Δεν θα πρέπει λοιπόν το 19,6 να το περικόψουμε ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να επιμείνει σε ένα 20% για μια μακροπρόθεσμη και άλλωστε αποδεδειγμένα αποτελεσματική στρατηγική. Ενώντα το επίπεδο το οποίο εμείς έχουμε επιλέξει για να έχουμε στο δυνατόν και οικονομική αλλά και αποτελεσματική διαχείριση των ε, δαπανών. Το 20% είναι το ελάχιστο απαραίτητο, πιστεύω. και δεδομένη τη ε, πολιτική ε, δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να κατέβουμε παρακάτω. Γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι πολύ θετική η προσέγγιση στις ε, διαπραγματεύσεις και για τον Brexit αλλά και εν ώψη των ευρωεκλογών. Θα έχουμε πολλά ζητήματα, βλέπουμε τις δυσκολίες ήδη με την Τουρκία, βλέπουμε τι δυσκολίε μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία και γενικά πολλά προβλήματα περί την Ευρώπη που αντιμετωπίζει και έλλειμμα υποστήριξη στις δημοκρατικές αρχές και αξίες και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια. για την ισότητα μεταχείριση των φύλων ήδη έχουμε κάνει επανειλημμένως ε, και δεκαετίες τώρα την ίδια συζήτηση. Εγώ θα πρότεινα η συμφωνία που έχουμε για την τρέχουσα θητεία να διατηρηθεί και σε αυτή τη συμφωνία. Για την προσεχή περίοδο, εάν να συζητηθεί κάτι, καλό θα ήταν να εισαχθεί η έννοια της εκούσιας προσπογραφής αυτούς τους κανόνες καθένα μπορεί να το προβάλλει αυτό στην προεκλογική του εκστρατεία, ότι τηρεί του κανόνε, ότι είναι διαφανή, ότι είναι υποδειγματικό κτλ. Επομένω και εκούσια προσωπογραφία, αλλά και κίνητρα. Νομίζω ότι θα είναι η πιο καλή λύση. Είναι και προ όφελο τη διαφάνεια, νομίζω, οι ίδιοι βουλευτέ να διαμορφώνουν τη διαφάνεια όπω θεωρούν ότι είναι πιο κατανοητή για τους πολίτες τους και πιο κατάλληλη για τη γραμματεία. Έχουμε δει πολλές νέες ε, προδιαγραφές το τελευταίο διάστημα. που μας επιβάλλουν πάρα πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο. Εγώ στο δικό μου το επιτελείο είχα έναν άνθρωπο που ασχολείται μόνο με τα λογιστικά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κοιτάξουμε. Και πρέπει να κοιτάξουμε και το κόστος που συνεπάγεται να έχουμε συνεργάτες ε, κατηρτισμένους, ε, τους βοηθούς μας που ταξιδεύουν στο Στρασβούργο κάθε φορά και αν δούμε τι είδους ε, επιβάρυνση σημαίνει αυτό γραφειοκρατική, διοικητική για το προσωπικό μας, θα ήταν καλό να μην είναι τόσο έντονη αυτή η διοικητική επιβάρυνση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αμοιβέ που δεν έχουν να κάνουν με εμά, αλλά με το προσωπικό μας. Και βέβαια αντίστοιχα θα πρέπει να δίνονται και οι αυξήσεις ε, αναλόγως ε, του κόστους και βεβαίως ε, αμοιβέ οι οποίες να ανταποκρινόνται στην ποιότητα και τη δουλειά των συνεργατών μας. Για τις εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι βάση της δημοκρατίας και το 2019 που κατά πόσο πιθανότητα μπορεί και να υλοποιηθεί το Brexit θα έχουμε και οι Βρετανοί συνάδελφοι αλλά και, και εμείς όλοι μια ιδιαίτερη δουλειά να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κατάλληλες λύσεις σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τους Βρετανούς συναδέλφους για να προσφέρουμε κατάλληλες λύσεις και για τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Μανκά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Άσουερθ με πολύ μεγάλη επάρκεια Νομίζω ότι και από τα σχόλια που άκουσα μέχρι τώρα θα στηρίξουμε τις προτάσεις του. Είχα θέσει κάποια ερωτήματα πέρυσι τον Απρίλιο Είχαμε πει ότι κάθε πέντε χρόνια θα προσπαθούμε όχι απλά να προσαρμόζουμε ε, από έτος σε έτος ανάλογα με τους δείκτες στον προϋπολογισμό, αλλά θα προσπαθούμε επίσης να εισάγουμε και νέες συγκεκριμένες θέσεις, έτσι ώστε κάθε πέντε χρόνια να έχουμε ένα πραγματικό προϋπολογισμό τον οποίο να προσαρμόζουμε ανάλογα με την εξέλιξη ε, για τα επόμενα τέσσερα. Νομίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και φοβάμαι ότι παρόλη την προσπάθεια την οποία πολλοί από μας ε, έχουμε κάνει δεν μας άκουσε η διοίκηση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ. Στο τέλος του χρόνου θα έχουμε ένα επιπλέον ποσό 7 εκατομμυρίων. Αυτό ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για θέματα επισκευών, κτηρίων κτλ. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε όμως το ποσό αυτό ε, για τις επιστροφές νωρίτερα και να προσπαθώσουμε έτσι να γλιτώσουμε ε, κάποιες καθυστερήσεις που θα οδηγήσουν σε επιβαρύνσεις λόγω των επιτοκίων των χρεών μας. Τώρα για, τις, για τα γραφεία ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διάφορες χώρες. Αυτό το οποίο εγώ διαπιστώνω είναι ότι υπάρχουν εννέα ε, γραφεία τα οποία είναι στη διάθεση των πολιτικών ομάδων και μπορούν να διατίθενται και να ενοικιάζονται στις πολιτικές ομάδες. Αυτό γίνεται σαν παράδειγμα στη Ρώμη. Ε, έχουμε στην ουσία χώρους ακίνητα στη διάθεσή μας, τα οποία δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε. Και μάλιστα οι μεγάλες πολιτικές ομάδες δεν γνωρίζουν πολλές φορές την δυνατότητα η οποία υπάρχει προς ενοικίαση των συγκεκριμένων χώρων που είναι διαθέσιμα στα γραφεία ενημέρωσης του Κοινοβουλίου στις διάφορες χώρες. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την δυνατότητα αυτή Αυτό είναι μια ιδέα την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε προσεκτικά εδώ και, αλλά και για αρκετό καιρό. Κύριε Τεπέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ήδη έχω πει ουσιαστικά στον κύριο Ashworth ότι είναι μια καλή έκθεση, ισορροπημένη, σωστά δομημένη και με σωστά επιχειρήματα και νομίζω ότι μιας και πρόκειται για ένα Βρετανό εισηγητή και μάλιστα των συντηρητικών ε, πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό. Πέραν τούτου θα ήθελα όμως να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς θα συμφωνήσω λέγοντας ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου δεν ε, φτάνει στο 20% που είναι ο κανόνας. Αλλά νομίζω επίσης ότι στην ουσία υπάρχουν κάποιες, ζητούνται κάποιες αυξήσεις δαπανών και δεν τις αναλύουμε σωστά αυτά τα αιτήματα. Βλέπουμε ότι χωρίς τις έκτακτες δαπάνες υπάρχει μια πραγματική αύξηση 3,26% σε σχέση με το 2017. 3,2% μπορεί να τεκμηριωθεί για θέματα προσωπικού, γιατί ακριβώς ε, εξεπλάγημεν όλοι από την προσαρμογή των μισθών με βάση το ισχύον σύστημα. Αλλά αυτό αφορά στο 68% των δαπανών. Ε, πρέπει να μου αποδείξετε ότι η σύνδεση με τις εξελίξεις των τιμών και με 2% δεν φτάνει κανείς το 3,26%. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι μισθοί που έχουν προκαλέσει αυτή την αύξηση. Εγώ έκανα εδώ και κάποιες ενδιαφέρουσες πράξεις. Προσπάθησα να δω τους τελευταίους χρόνους ε, ποιες ήταν οι θέσεις του προϋπολογισμού οι οποίες συστηματικά ήταν υπερεκτιμημένες όπου τα τελευταία χρόνια υπήρχε λοιπόν ε, να, η δυνατότητα να διαπιστώνουμε ότι από κάποιες γραμμές παίρναμε στο τέλος του χρόνου χρήματα για να χρηματοδοτούμε τις υπόλοιπες. Αυτό γίνεται με πολύ τακτικό θα έλεγα χαρακτήρα και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Ταυτόχρονα μας λένε ότι οι πιστώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την χρηματοδότηση του κτηρίου Κάντα. Το κτίριο Κάντα στις προβλέψεις δαπανών για τον επόμενο χρόνο ε, περίπου απαιτεί 60 εκατομμύρια. Αν λάβω υπόψη τις δαπάνες που ήδη έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, ήδη για την ολοκλήρωση του κτηρίου Αντενάουερ υπάρχουν 33 εκατομμύρια επιπλέον. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να βρούμε 27 εκατομμύρια από το λεγόμενο ραμασάζ στο τέλος του χρόνου, το οποίο είναι σε ετήσια βάση από 50 με 70 εκατομμύρια. Λοιπόν, πρέπει να τα δούμε λίγο πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Ρούμπιχ, ο οποίος λέγει ότι οι δαπάνες αυτές είναι καλοδεχούμενες. Πλησιάζουμε σε εκλογές και η στρατηγική αυτή δεν είναι η ορθή. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει κάποια χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού και κάποιες αιτήσει αύξησης των δαπανών να τα επανεξετάσουμε. Τώρα για την ασφάλεια και την ασφάλεια. Κοιτάξτε, εδώ ε, να πούμε ότι 25 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όπως είπε ο κύριος Ashworth, περιλαμβάνονται στις έκτακτες δαπάνες, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, δεν πρέπει να είναι στις έκτακτες πιστώσεις και δεν νομίζω ότι η προστιθέμενη αξία των 25 εκατομμυρίων ευρώ είναι υψηλότερη από το σύνολο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των δημοσιεύσεων, στον τομέα της ενημέρωσης κτλ. Η προσπάθεια στην οποία γίνεται είναι να πείσουμε τους πεπισμένους. Ε, δεν είναι αυτό ενδιαφέρον. Το θέμα είναι να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον αυτών που έχουν διαφορετική άποψη και αυτών που είναι ξεκάθαρα εχθρικοί απέναντι στο Κοινοβούλιο και στην Ένωση. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δούμε λίγο ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι μέσω του προϋπολογισμού αυτού. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ε, εκτιμώ ιδιαίτερο τις παρατηρήσεις του Ashworth όταν ασκεί κριτική ε, στις 76 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου ε, συμφωνώ επίσης με αυτό το οποίο είπε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε κάποιες δαπάνες στον τομέα των πολιτικών ομάδων και των πολιτικών ιδρυμάτων και μάλιστα πάνω από τον δίκτυ τιμών και νομίζω επίσης ότι είναι ευαίσθητο βέβαια το θέμα της αποζημίωσης γενικών εξόδων. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση την οποία κάνει ε, είναι να ζητήσουμε από το Προεδρείο και από τον Γενικό Γραμματέα να αναθεωρήσουν, να μεταρρυθμίσουν πλήρως το σύστημα το οποίο από την επόμενη περίοδο ε, θα πρέπει να λειτουργήσει. Αν κάνουμε κάτι τώρα θα είναι βιαστικό, θα είναι απροπαρασκεύαστο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε τις ε, δαπάνες για γενικά έξοδα τις αποζημιώσεις για γενικά έξοδα από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο και πάνω σε αυτό πρέπει ο Γενικός Γραμματέας και το Προεδρείο να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Ντενανό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ο συνάδελφος Μάνκα και άλλοι συνάδελφοι, Είμαι υπέρ του να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιστώσεις. Και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η εισηγητής λέει ότι θα πρέπει καταρχάς και κατά προτεραιότητα να ασκεί τις συνομοθετικές του αρμοδιότητες αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε μια φούσκα απομονωμένη. Θα πρέπει να επικοινωνούμε για να το πετύχουμε. Πρέπει να ανοίξουμε προς τα έξω, να γνωστοποιούμε το ποιες είναι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι τα βραβεία που δίνουμε σε διάφορους τομείς δείχνουν κάποια πράγματα όπως το Λουξ για τον κινηματογράφο που προωθεί κινηματογραφικές δραστηριότητες που βασίζονται στις κοινωνικές συνθήκες που σοβούν στην Ευρώπη σήμερα. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε το χώρο αποκλειστικά στη διάθεση της Επιτροπής και στο Συμβούλιο. Μένουμε πάντα κάτω από το 20% και νομίζω ότι τα περιθώρια όποια και αν είναι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να γνωστοποιηθεί η σημασία και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σημασία την οποία θα πρέπει να δίνουν οι πολίτες έτσι ώστε να πάρουν μέρος στις ευρωεκλογές. Συνεπώς λοιπόν έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε στον κόσμο καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να τους πείσουμε να προσέλθουν στις κάλπες. Κυρία Γουαρδιαζάβαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποια γενικά σχόλια, αν και πολλά υπόθηκαν από τους δύο προηγούμενους συναδέλφους. Εμείς συμμεριζόμεθα με πολλές από τις βασικές αρχές τις οποίες εξέφρασε ο κύριος Ashworth, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μεγάλη φροντίδα για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται το δημόσιο χρήμα και θα πρέπει τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας να τα χρησιμοποιούμε κυρίως για να εξηγούμε με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι τώρα τις δράσεις μας. Και επίσης συμφωνώ με αυτά τα οποία υπόθηκαν για κάποιες ε, επαναληπτικές χρόνο με χρόνο ε, καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται και οι οποίες χρήζουν επανεξέταση. Είναι λογική λοιπόν την οποία λέει ο κύριος Άσχορθ, η πρόταση του κύριου Άσχορθ, έτσι ώστε το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας να μας κάνουν μια ξεκάθαρη πρόταση, πολύ συγκεκριμένη, την οποία στον τομέα των αποζημιώσεων για τα γενικά έξοδα των βουλευτών, σαν παράδειγμα, να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή από, τον επόμενο, από την επόμενη εκλογική περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε την καλύτερη χρήση του δημοσίου χρήματος και ταυτόχρονα να υπερασπιστούμε την χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Μιας όσοι είμαστε φιλοευρωπαίοι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες και οι διαδικασίες που οδηγούν σε αυτό θα πρέπει να περνούν και μέσα από τις πολιτικές ομάδες και την ενίσχυσή τους και θα πρέπει τα πολιτικά ευρωπαϊκά κόμματα να μην είναι ένα απλό σύνολο 27 ή λιγότερων χωρών, αλλά να περάσουμε σε ένα πραγματικό εξευρωπαϊσμό της πολιτικής κοινής. Τώρα για τις διάφορες μελέτες τις οποίες παραγγέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά, τις μελέτες αυτές και τις έρευνες, εμείς δεν λέμε ότι αμφισβητούμε την, την ποιότητα των συγκεκριμένων προτάσεων, αλλά λέμε ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε επικαλύψεις και θα πρέπει να μην κάνουμε δύο φορές, ε, να μην προσφεύγουμε δύο φορές σε υπεργολαβικές ε, δραστηριότητες. Τώρα για τον πληθωρισμό. Πολλές ε, γραμμές του προϋπολογισμού έχουν αυξηθεί λόγω του πληθωρισμού και στα πλαίσια της αύξησης των μισθών των εργαζομένων Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να αυξηθεί λίγο ο προϋπολογισμός ε, λόγω ακριβώς και της αύξησης του πληθωρισμού πλέον, αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε αν αυτή η διαφορά, αυτή η αύξηση ανταποκρίνεται μόνο σε αυτό ή και σε κάτι περισσότερο. Τώρα για τα βραβεία τα οποία δίδουμε σε ετήσια βάση, όπως το βραβείο για τον κινηματογράφο, το βραβείο Λούξ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε μέχρι τώρα γιατί είναι χρήσιμη. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι κάνει δύο προτάσεις ο κύριος Άσχουαρθ. Ζητά την ενίσχυση του διαλόγου σαν παράδειγμα με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους τομείς ή σε συγκεκριμένους μάλλον τομείς. Και μια άλλη ιδέα είναι τα χρήματα τα οποία προορίζονται για την προεκλογική εκστρατεία. Νομίζω ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να έχουν σαν βασικό στόχο το να εξηγούν τι, τον ρόλο, την ουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εκλογικό σώμα. Όχι να χρηματοδοτούν γενικά τις δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων. Απλά θα πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να επισημάνουμε το ποιε είναι οι δυνατότητες χρήσης των πιστώσεων για την προεκλογική εκστρατεία καλύτερα. Ο κύριος Τάραντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι με ικανοποιεί ιδιαίτερα το ότι έχει προχωρήσει τόσο καλά το κείμενο στην αποτελευταία μας συνεδρίαση ούτως ή άλλως αποτελούσε εξαίρετη βάση συζήτηση. Και με το κείμενο που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που εισήγαγε ένα σχόλιο της τελευταίας συνεδρίασης για το η διάρκεια ζωής του κτηρίου Πολών Ρισπακ και τα λοιπά σχόλια για την ε, κτηριακή πολιτική για τις οικονομίες. Είναι απόλυτο φυσιολογικό να βγουν οι επεξηγήσεις ψήφου από τις ώρες μεγάλης ακρόασης όπως θα τις λέγαμε και να πάνε στις ε, μέσονίκτιε συνεδριάσεις και θα έλεγα ακόμα και να γίνονται μόνο γραπτός και να μην μεταφράζονται. Ακόμα καλύτερα αλλά δεν ξέρω αν αυτό ξεπερνά τα όρια ενός, ε, μιας εκθέσεως του προϋπολογισμού για αν διαφωνούν κάποιοι άλλοι. Εάν θέλουμε να δώσουμε χρήματα για το πρόγραμμα το προεκλογικό για την ενημέρωση για τις εκλογές, με εκπλήσει το γεγονός ότι η κυρία Γκάρδια Ζαβάλ βλέπει υπερβολικά πολλούς περιορισμούς στην ιδέα αυτή γιατί θα θυμάστε ότι είχαμε ζητήσει να συμμετέχει στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή ο εκπρόσωπός μας, αλλά ο Γενικός Γραμματέας δεν είχε δώσει σαφή απάντηση για το αν θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Δεν το είπε ρητά. Εάν ήταν παρόν λοιπόν δικός μας ε, συνάδελφος, ίσω να ήταν λιγότεροι περιορισμοί. Άπαξ όμως και δεν συμμετέχει στι προπαρασκευαστικές εργασίε η Επιτροπή των Προπολογισμών, θα πρέπει να έχουμε κάποιου αυστηρούς περιορισμού αυτά και θα ήθελα επίση να συμπληρώσω ότι ίσως η δημοσιονομική διαδικασία, η διαδικασία για τον προϋπολογισμό φέτος ε, να φανεί λιγότερο ε, τεταραγμένη. Αυτό οφείλεται και βέβαια στον εισηγητή και την καλή διάθεση. Γι' αυτό και λυπούμε που αποχωρούν οι Βρετανοί. Ο πρόεδρος. Ναι είναι η ώρα της συγκίνησης. Ο κύριος Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή. Με ικανοποίησαν ιδιαίτερα κάποιες από τις προσθήκες που έκανε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Ήταν καλή και η πρόταση για την εξέταση της αναθεώρησης σε όρους διαφάνειας των γενικών ε, δαπανών των βουλευτών. Πρέπει δηλαδή να δοθεί και η συνέχεια στα όσα είχε ψηφίσει κατά δύο φορές τουλάχιστον νομίζω η Ολομέλεια προς το στόχο της διαφάνειας. Άρα και εδώ θα ήταν καλό να έχουμε μάλιστα μια καθοδήγηση από τη Γενική Γραμματεία για ένα κείμενο, μια πρόταση αναθεώρησης προς το στόχο της διαφάνειας των δαπανών. Ως ομάδα είμαστε κατά της ενίσχυσης των δαπανών του προπολογισμού. Είναι πολλέ οι περικοπέ που κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των σχεδόν εισηγητών θα σα προτείνω. Γραμμικέ περικοπέ, μπορούμε να τι συζητήσουμε στα διάφορα κεφάλαια και ίσω αυτή η αύξηση του 3,26% που μάλλον είναι υψηλή δεδομένης της κατάστασης και τη γενική ανάπτυξη στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται μάλλον υψηλό ποσοστό, θα πρέπει λοιπόν να το ξανασυζητήσουμε. Ας είμαστε προσεκτικοί για το δίκτυο αυτό, γιατί αφορά και τους ε, μισθούς και την ε, ε, διεύρυνση με τις 12 χώρες και άλλωστε είναι και γενικοί δίκτες αυτοί, δεν αφορούν μόνο δηλαδή πρώτες ύλες και δίκτυοι καταναλωτή δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονό ότι πολλέ χώρε είναι σε αποπληθωρισμό. Αν ακολουθήσουμε δίκτυο πληθωριστικό, θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένα ε, καλάθι για τον προπολογισμό και όχι γενικού όρου και ποσοστά. Σε προηγούμενε εκθέσει σχετικέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ήδη εκφράσει τι θέσει μα. Ε, θα θέλαμε να μειώνονται μάλλον οι δαπάνε για να πάνε προς ε, τον εκδιδενισμό. Για την εκστρατεία την προεκλογική του 2019, 25 εκατομμύρια, που άλλωστε μας είχε δώσει και κάποιες ενδείξει στην προηγούμενη συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας για το πώς θα δαπανηθούν τα ποσά αυτά, αλλά εμείς διαφωνούμε ως προς την χρήση των κονδύλων αυτών, γιατί και σε σχέση με την ε, εκστρατεία του 2014, την προεκλογική, δεν είδαμε πολύ καλά αποτελέσματα η συμμετοχή. Σε σχέση με τις εκλογές του 2009 είχε μειωθεί σημαντικά το 2014, αλλά δεν έφεραν αποτελέσματα αυτές οι ταπάνες. Για τις μελέτες, ε, τις σχετικές με την ανακαίνιση του PHS και τα 14 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται, πάλι πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια δαπάνη υπερβολική όπως άλλωστε σημείωσαν και άλλες ομάδες και ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Αυτά για την ε, σύγκριση με το παρελθόν πρέπει να πω ότι είχαμε εξαίρετους ε, ε, συντάκτες εκθέσεων. Φέτος είναι ακόμη πιο φιλόδοξη η έκθεση, μια πολύ καλή βάση εργασίας και συνεργασίας και πιστεύω θα μας οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι άλλωστε θα δώσει ένα ψημα και στους και να προσφέρουν με τις ιδέες τους ακόμη περισσότερο στη βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ. Κύριε Μιάντο. Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι σύντομη. το συγγνώμη γιατί ο σκιώδης ε, και ο Σούμερη ζητάει συγγνώμη. Σε γενικέ γραμμέ, συμφωνούμε με τις προτεραιότητες ε, του εισηγητή και με αρκετά ε, από τα προβλήματα που έθιξε. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερη λογοδοσία για τις κοινωνικές πτυχές ε, και το προσωπικό και για όσους επηρεάζονται άμεσα από τις συμβάσεις με τρίτους, ε, ειδικά επίσης θετικά τα βήματα για την διαφάνεια, ειδικά η προτάση του κυρίου Μάνκε και νομίζω ότι είναι θετικό το ότι αναγνωρίζεται η Ιρλανδική γλώσσα Μιλάμε για προσβασιμότητα από τους ε, πολίτες και επικοινωνία μαζί τους ε, και το ότι σεβόμαστε όχι μόνο την Ιρλανδική γλώσσα, αλλά στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι σεβόμαστε την πολυγλωσία και τους ε, πολιτισμούς και βεβαίω αναμένουμε και την δυνατότητα να μπορέσω και εγώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα πριν από το τέλος της θητείας. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει τον λόγο. Θα ήθελα... Και θα ήθελα και προσωπικά να συμφωνήσω στους επένους προς τον εισηγητή μας. Ήταν ε, ιδιαίτερα ε, ενημερωτικές οι εξηγήσεις. για το 20% του πέμπτου τίτλου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουμε μια κάποια σύνεση, διότι εάν οι λοιπές πάνω στο τίτλου 5 αυξάνονταν σημαντικά, καλό θα ήταν να μην επιδιώκουμε να διατηρούμε το 20% ε, πάντοτε, διότι αυτό δεν θα σήμαινε βέβαια χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων. Η Ευρώπη κάθε χρόνο απευθύνει συστάσεις στα κράτη-μέλη να δείξουν λιτότητα και πειθαρχία στη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Ε, τι θα γινόταν το κύρος του Κοινοβουλίου, αν το ίδιο αυτό αύξανε κατά 3,26 τις, τις δημοσιονομικές του δαπάνες. Αντίφαση θα ήταν βέβαια. Πάντως η νομική βάση που ορίστηκε πριν από τρία χρόνια λαμβάνει υπόψη της αυξήσεις των μισθών σε διαφορετικές χώρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο αντιμετωπίζουν κόστος ζωής αντίστοιχο με αυτό της Βαρσοβίας ή άλλων κρατών. Ας προσέχουμε λοιπόν γιατί μπορεί να έχει στρεβλωτικό αποτέλεσμα αυτός ο δείκτης. Και αν η κοινή γνώμη λαμβάνει γνώση των μηχανισμών αυτών θα μπορούσε και να αμφισβητήσει τη βασιμότητά τους. Γιατί το θέμα δεν είναι να χρησιμοποιούμε 25 εκατομμύρια για την ε, ε, επικοινωνιακή πολιτική που θα αποδείξει την προσθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή των Προπολογισμών σαν κύριο και πρώτο καθήκον έχει να επιδείξει πνεύμα πειθαρχία και λιτότητα και εγώ εκ πρώτη όψεω πρέπει να πω ότι αισθάνομαι δυσφορία γιατί βρισκόμαστε μέσα σε ένα μηχανισμό ο οποίο ε, θέτει σε κίνηση ένα μηχανισμό δαπανών σε συνθήκες που μπορεί να είναι και αμφισβητήσιμες και ε, αντικείμενο επικρίσεων. Βλέπουμε βέβαια κάθε φορά και χάρη στους εισηγητές μας ε, ξεκάθαρα με βάση τα έγγραφα ποια είναι η κατάσταση, όμως για τα κτίρια και για τις προοπτικές της, ε, της κτηριακής πολιτικής δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Το να κάνουμε λοιπόν μια σόρευση των πόρων, ουσιαστικά, μια σάρωση μάλλον των πόρων, ουσιαστικά ανατρέπει το νόημα του προπολογισμού, διότι αναλαμβάνουμε υποχρεώσει δαπανών, ξέρω ότι τελικά θα μα κοστίσουν τα διπλώσια και χωρίς να έχουν καλυφθεί τα έξοδα από άλλου πόρους. Και γι' αυτό θα ήθελα προσωπικώ να πω ότι δεν αισθάνομαι ικανοποίηση από την εικόνα αυτή και να πω ότι επίση θεωρώ πω για τι επενδύσει έχουμε ακόμα σημαντικό περιθώριο βελτίωση. Δίνω ωστόσο το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ελιάνη, θέλω να ευχαριστώ τους συναδέλφους και για τα καλά τους λόγια, αλλά και για τις επικοδομητικές τους παρατηρήσεις. Για το τελευταίο σχόλιο, τα τελευταία λόγια του Προέδρου, ναι, το 20% είναι κατευθυντήρια γραμμή για τα κονδύλια που πρόκειται να δαπανίσουμε, αλλά θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η σημασία δεν έχει το ποσό, αλλά το τι το κάνουμε το ποσό αυτό, εάν δηλαδή φέρνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα η δαπάνη. Και εδώ αισθάνομαι ικανοποίηση σε σχέση με τα σχόλια των συναδέλφων, διότι βλέπουμε σαν πάγια εποδό την πειθαρχία πρώτον, τη διαφάνεια δεύτερον και την λογοδοσία τρίτον. εποδό την οποία και εγώ θα ήθελα να ελπίζω ότι βλέπετε σε όλη μου την έκθεση. Για το GA ιδιαίτερα αλλά γενικότερα για τις ομάδες και τα ιδρύματα είναι κάτι το οποίο όπως είπε και ο θα πρέπει να μας απασχολήσει για την προσεχή θητεία. Δεν προλαβαίνουμε στην τρέχουσα θητεία να το κλείσουμε το θέμα αλλά πρέπει ως Επιτροπή να προβούμε στα απαραίτητα βήματα ώστε να καθοδηγήσουμε το Προεδρείο για την ε, εγκαθίδρυση μιας βέλτιστης πρακτικής ε, που θα πρέπει συνέχεια να γίνει μια ε, κοινή πρακτική για όλους. Για τα σχόλια του Παουλ Ρούμπιχ, τα έξοδα γραμματείας. Εμένα με ανησυχεί όχι το ύψος των δαπανών εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά το επίπεδο των δαπανών στις λεγόμενες αποζημιώσεις γραμματείας στις χώρες προελεύσεως. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, μυρίζουμε τα σχόλια των, ε, του Πρόεδρου και του κυρίου Ντεπρέ σε σχέση με τη σάρωση των δαπανών. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια. Οι συνάδελφοι έκαναν λόγο για τις ε, δαπάνες και το κόστος της προεκλογικής εκστρατεία και ιδιαίτερα στις δύο παρατηρήσεις και ερωτήσεις της Άιντα ε, για το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα προγράμματα ε, επικοινωνίας. Ταυτόχρονα θα δώσω την απάντηση στις δύο ερωτήσεις. Πρώτο σκέλος, θέλω σαφήνεια, θέλω να ξέρουμε τι κάνουμε. Και αυτό ως προσωπική παρατήρηση και κατόπιν βέβαια και τη εμπειρία τη εκστρατεία για το δημοψήφισμα στη χώρα μου, η έλλειψη πληροφορία στη χώρα μου, και δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν είναι αντίστοιχη η έλλειψη πληροφορία στα λοιπά κράτη, αλλά και σε σχέση με το Κοινοβούλιο, είναι πολύ ανησυχητική. Δεν ε, είναι ρόλο του Κοινοβουλίου ασφαλώ να ξεκινήσει ένα πόλεμο προεκλογικής προπαγάνδα. δεν θα το έλεγα έτσι, θα ήταν κάτι το εσφαλμένο άλλωστε, αλλά είναι καλό να προβάλλεται αυτό που πράττει το Κοινοβούλιο, γιατί έχει σημαντικό ρόλο. Και εδώ επανέρχομαι σε μια παρατήρηση που έκανα νωρίτερα. Γιατί αυτό θα πρέπει να το δούμε σε μια έκτακτη δαπάνη για ένα έτος εκλογών. Πρέπει να είναι δαπάνη πάγια και δραστηριότητα πάγια. Γι' αυτό θα ήθελα μια πιο ομαλή κατανομή της δαπάνης. Επίσης ευχαριστώ και τον κύριο Ταράντ και τον κύριο Ντεπρέ για τα σχόλια. Εν γέννη ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, την κυρία Νιριάντα Άντα και και Σμίλια Φάρτσα. Thank you, Chairman. And to think that an Englishman is giving an Irishwoman back her language, that's an extra... Να και ο Βρετανός ο οποίος επιστρέφει τη γλώσσα της στην ε, Ιρλανδή. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Bien, donc, vous aurez une réunion avec euh, les... Καλώς λοιπόν, συνεδρίαση προβλέπεται με τους σκιώδεις ηγητές στις προσεχείς ημέρες. Επισημαίνω ότι οι τροπολογίες για το σχέδιο εκθέσεως του κ. Άσχουρεθ θα κατηθούν έως τις 15 Μαρτίου, μία το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 3 Απριλίου. Στην Ολομέλεια, από ό,τι βλέπουμε, θα πάει η ψηφοφορία της έκθεσης ή στις 5 ή στις 6 Απριλίου. Και τώρα θα δούμε τα πιλωτικά έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Δύο είναι οι εισηγητές, ο κύριος Μούρεσαν, γενικός εισηγητής για το 2018 και ο κύριος Γκάιερ, τον οποίο αντικαθιστά η κυρία Γκαρδιάζα Πάλεν προκειμένου. Ποιος ξεκινάει, ο κύριος Μουρεσάν, ο κυρία Γκαρδιάζα Πάλεν. Ο κύριος Μουρεσάν, νομίζω είναι καλύτερο να ξεκινήσει η συνάδελφος γιατί ο Γιάννης Καΐρ είναι αρμόδιο για φέτο, ενώ εγώ θα έχω την επόμενη χρονιά το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορώ να είμαι νομίζω σύντομη. Μου ζητήθηκε να μεταφέρω κάποιες απόψεις του εισηγητή. Πρόκειται για μια ενδιάμεση ουσιαστικά προσωρινή έκθεση αν θέλετε λειτουργεί ενημερωτικά περισσότερο σε σχέση με τα πιλωτικά και προπαρασκευαστικά προγράμματα από τα 79 τα οποία εγκρίναμε τα περισσότερα έχουν ξεκινήσει αλλά πέντε από αυτά ε, στα πλαίσια της κάρτας εκτέλεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστικά έλλειψη της νομικής βάσης και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει επανεξέταση των θεμάτων αυτών και μάλιστα κάποια από αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ευαισθησίας. Για τα υπόλοιπα τώρα υπάρχουν άλλα τέσσερα από τα προγράμματα αυτά. Έχει υπάρξει μια προκαταρτική έκθεση από πλευράς της Επιτροπής η οποία αναζητεί ε, τρόπους ε, με τους οποίους να μπορέσει να τα εφαρμόσει. Ακόμα όμως δεν έχει προχωρήσει σε αυτό. Δεν ξέρω αν εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει λίγα περισσότερα στοιχεία για την φύση του προβλήματος τα οποία, ε, των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει σε σχέση με τα τέσσερα αυτά στα οποία βρίσκεται ακόμα σε προκαταρτική φάση. Τώρα δεν ξέρω τι περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορούσα να πω που περιλαμβάνονται σε αυτήν την προκαταρκτική έκθεση. Έτσι και αλλιώ θα ασχοληθούν με αυτά οι επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες τομεακά τις καλύπτουν. Ο κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγητής ε, του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι οπωσδήποτε κάθε βουλευτής ε, μπορεί να καταθέσει προτάσεις για πιλωτικά έργα και παρασκευαστικές δράσεις και το πρώτο στοιχείο που είναι σημαντικό για να υποβληθεί μια τέτοια πρόταση η οποία θα είναι επιτυχής ε, στην αξιολόγηση και θα αρχίσει να εφαρμόζεται είναι ότι όλα τα πιλωτικά έργα θα πρέπει να αποσταλούν σε μια προαξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις 3 Μαΐου. Οπότε 3 ε, Μαΐου η προθεσμία για την προαξιολόγηση της ε, Κομισιόν και να πω στους συναδέλφους πως ακόμα και τα υφιστάμενα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις που θα παραταθούν πρέπει να πάνε στην προαξιολόγηση της Κομισιόν. Μετά η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τα ευρήματά της και μετά πρέπει οι συνάδελφοι να γνωρίζουν το ότι κάθε πιλωτικό έργο υπερπαρασκευαστική δράση πρέπει να κατατεθεί ως τροπολογία στον προπολογισμό του επόμενου έτους και οι προθεσμίες είναι 31 Αυγούστου για τροπολογίες από επιτροπές ή βουλευτές και 7 Σεπτεμβρίου για τροπολογίες ε, των ε, πολιτικών ομάδων. Και μετά το φθινόπωρο θα ετοιμάσουμε ένα πακέτο όπως έγινε και πέρσι και βεβαίως θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πιλωτικά εκείνα έργα οι προπαρασκευαστικές δράσεις που έχουν λάβει θετική προαξιολόγηση από την Κομισιόν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τα ξέρουμε αυτά μέχρι τις 3 Μαΐου και ειδικά όσα έλαβαν βαθμό α ή αβ από την Κομισιόν. Και να πω πως ε, όταν παρουσίασα το σχέδιο έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές του προπολογισμού για το επόμενο έτος, είπα πως οι προτεραιότητες του προπολογισμού για το επόμενο έτος θα είναι ανάπτυξη, οι δουλειές και η ασφάλεια των πολιτών. Ανάπτυξη και δουλειές γιατί αυτό ε, ζητάνε οι πολίτες της Ευρώπης να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση που οδηγεί σε δημιουργία θέσεων εργασία, σε καινοτομία, σε υποδομές. Ε, θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, θα στηρίξουμε τους νέους, ειδικά τους νέους επιχειρηματίες και όλα αυτά θα επιτύχουν βεβαίως μόνο εάν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αυτό είναι σημαντική και η ασφάλεια. Θα στηρίξουμε τις υπηρεσίε εκείνες τη Ένωση που εργάζονται στον τομέα τη δικαιοσύνης και εσωτερικών και επειδή αυτές θα είναι οι βασικές προτεραιότητες του προπλογισμού για το επόμενο έτος, θα δοθεί ειδικό βάρος στα πιλωτικά έργα σε αυτές τις ε, κατευθύνσεις. Τούτων λεχθέντων, θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε και αναμένω ενδιαφέροντα πιλωτικά έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις που θα προτείνουν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ και εισηγητά. Ίσως η Κομισιόν που εκπροσωπείται από τον κύριο Γιώχαν Ιρελ... Α, ο κύριος Ντορνάλτο πρώτα, συγγνώμη. Ναι, ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, λέει ο κύριος Ντενάντο. Κοιτάξτε... Η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας έχει, είναι αυτό το θέμα. Είχαμε ξεκινήσει από το 2015, έκτοτε δεν ακούσαμε τίποτα από την Επιτροπή και θέλω να μάθω επιτέλους εάν θα υπάρξει κάποιο έργο, αν θα κατεθεί κατά κάποια πρόταση για να δοθούν απαντήσεις. 700 συν 200.000 ευρώ, 900 το όλων, ελπίζω να διατηρηθούν για τη φετινή χρονιά. Ευχαριστώ. Κύριε Ναβακοφ, ναι και εγώ έχω μια παρατήρηση για τα πιλωτικά έργα. Ορισμένα πάνε πολύ καλά βεβαίως, ε, πολλά όμως δεν έχουν περιγραφεί με περισσότερες λεπτομέρειες. Πολλές φορές ε, ζητούμε πληροφορίες από την Επιτροπή και οι εκπρόσωποι της μας λένε «Α, όλα πάνε καλά». Αλλά εμείς που υποστηρίξαμε αυτά τα πιλωτικά έργα δεν λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες. Και σας λέω ξεκάθαρα ότι με ενδιαφέρει πώς υλοποιείται, όχι οι λεπτομέρειες, με ενδιαφέρει πώς υλοποιείται ένα έργο από την Επιτροπή. Και να δούμε ότι πράγματι αυτό είναι το έργο το οποίο υποστηρίξαμε. Χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, μας έδωσε τις προτεραιότητες ο Γενικός Εισηγητής για να κάνουμε τη διάκριση και την επιλογή μεταξύ των διαφόρων πιλωτικών έργων. Να βάλουμε και την επικοινωνία εκεί μέσα. Μια και νωρίτερα μιλούσαμε για το ζήτημα της επικοινωνίας, της επικοινωνικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκέφτομαι πολλές φορές ότι οι δημοσιογράφοι πολλές φορές μας προσεγγίσουν ε, αναχώρα, ως εκπρόσωποι χώρας. Αν είχαμε ένα είδος εράσμου των νέων ε, δημοσιογράφων, να τους βοηθήσουμε δηλαδή να επικοινωνούμε δημοσιογράφους άλλων κρατών, ίσως αυτό να ε, ενίσχυε και το ενδιαφέρον τους και ίσως να βελτίωνε και την επικοινωνιακή μας ε, πολιτική και την παρουσία μας, ε, τον τρόπο με τον οποίο διάφορες ε, αρχισυνταξίες των εφημερίδων δίνουν χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη σημερινή εικόνα. Κύριος Γιώχαν Γκιούρερ εντωμεταξύ, εκ μέρους Τι γίνεται. Πώς αξιολογούνται τα έργα, πώς ταξινομούνται αυτά ως α, β, γ, δ. Περιμένουμε τα φώτα σας και βέβαια πώς μπορούμε να λαμβάνουμε πιο σαφείς πληροφορίες, ώστε εκείνοι που προάγουν, που προβάλλουν, που υποστηρίζουν τα πιλωτικά έργα να έχουν και την εικόνα της υλοποίηση τους μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω, καλώς ορίζουμε τη σημερινή συζήτηση και θα θέλαμε να επαναλάβουμε και να τονίσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 79 Πολιτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων εφαρμόζονται 70 από τα 79 τέσσερα αναλύονται ακόμα από την Κομισιόν και για να απαντήσω στο ερώτημα του εισηγητή μπορώ να πω ότι δεν έχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες καθώς η έκθεση δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα οπότε για τα τέσσερα επιπρόσθετα έργα δεν έχω άλλες ε, πληροφορίες, αλλά απριόρι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλά ακόμα τα μελετάμε και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής, οπότε ελπίζω να έχουμε καλά νέα και για τα τέσσερα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Οπότε μένουν πέντε ακόμα πιλωτικά έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό το είχαμε πει ήδη στο, στην επιστολή της Κομισιόν της 26ης Οκτωβρίου γιατί καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομική βάση και όπως συμφωνήσαμε στο κοινό κείμενο για τον προπολογισμό του 2017 όπου δυνατόν η Κομισιόν θα μεταφέρει τα κονδύλια στην ανάλογη νομική βάση που καλύπτει αυτές τις ε, πρωτοβουλίες μόνο εάν είχε ψηφιστεί υπό διαφορετικό τίτλο του πολιτικού δημοσιονομικού προγράμματος ε, ε, από την νομική βάση μόνο τότε δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα κονδύλια. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στον ε, εισηγητή για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που προτείνει. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να κάνει την αξιολόγηση εγκαίρως πριν από τον τριμερή διάλογο του καλοκαιριού και εγκαίρως ε, για να γίνουν οι διαβουλεύσεις και στις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Για τα συγκεκριμένα ερωτήματα των βουλευτών για ένα συγκεκριμένο έργο πιλωτικό ε, θα πρέπει να επανέλθω γραπτός. Δεν έχω συγκεκριμένες πληροφορίες αυτή τη στιγμή για την καλύτερη ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Προφανώς είμαστε στην διάθεσή σας, αλλά είχαμε την εντύπωση ότι η έκθεση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα παρέχει σημαντικές πληροφορίες και ουσιαστικές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, Κύριε Σιγητρία εκτιμάτε ότι οι απαντήσεις ε, της Κομισιόν απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ούτως ή άλλως είναι συμπληρωματικές. Ο κύριος Μουρεσάνη είπε ότι ε, στις 3 ε, Μαΐου 12 η ώρα είναι η προθεσμία για τα πιλωτικά αυτά έργα τα οποία θα πρέπει να προαξιολογηθούν πριν περάσουμε στα επόμενα θέματα. Λοιπόν, Έχουμε τώρα, όπως είπαμε, το σχέδιο γνωμοδότησης για την προώθηση, προαγωγή της σύνδεσης στο διαδίκτυο στις τοπικές ε, κοινότητες. Ε, Κυρία Νηριάντα, είστε έτοιμοι? Ναι. Βεβαίως. ιδιαίτερα στο τέλος μια συνεδρίαση στη Δευτέρα το απόγευμα. Είναι μια απλή ιδέα. Ο βασικός στόχος είναι να προσπαθήσουμε να εξοπλίσουμε τα περισσότερα χωριά της Ευρώπης και της πόλης με ελεύθερη δωρεάν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Δεν απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα. 120 εκατομμύρια από το 17 μέχρι και το 19 για την εγκατάσταση των συστημάτων Wi-Fi. Ε, οι μηχανισμοί θα εγκαθίστανται σε δημόσιους χώρους, ε, πάρκινγκ, ε, μουσεία, κοινή ωφέλεια κτίρια γενικότερα. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε γεωγραφικά τις περιφέρειες με ισορροπημένο τρόπο. Θα διευκολύνουμε κυρίως φυσικά τις κοινότητες οι οποίες δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό θα βοηθήσει επίσης τις ε, μικρές περιοχές, τις απομονωμένες περιοχές. Σε κοινωνικό επίπεδο θα είναι ωφέλιμο. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να διαφωνήσει. Θα βοηθήσει την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τον ηλεκτρονικό ε, τουρισμό επίσης Νομίζω ότι οι περιφερειακές ζώνες της Ευρώπης, αυτές οι οποίες είναι μακράν των μεγάλων πόλεων, στις οποίες υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες σύνδεσης, ε, θα ωφεληθούν από αυτό. ...20.000 σαν μεμονωμένη τέτοια μονάδα Wi-Fi. Οι διαδικασίες δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικές. Ε, μπορεί να υπάρξουν online ε, αιτήσει για την σε αυτές. Δεν νομίζω ότι περισσότερες λεπτομέρειες χρειάζεται να δώσουμε τώρα. Είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει σαφώς τη συνδεσιμότητα των περιφερειών και οι απόψεις μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα θετικές. Αν έχετε κάποιες επιμέρους ε, προτάσεις στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας έκθεση. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακόμα και αν η συγγήτρια λέει ότι δεν υπάρχουν ζητήματα, εγώ έχω κάποια θέματα με τέτοια έργα και να σας πω γιατί. Είναι κάποιο δουλικότητα από την πλευρά της Κομισιόν ή σαν να ρίχνουμε φιστίκια στα ζώα στο ζωολογικό κήπο και δεν βοηθάει πάντα. Οπότε υπάρχει μια, μια λέξη ε, στα αγγλικά που περιγράφει την κατάσταση. απερχιωμένος λέμε ε, και υπάρχει και ένα άλλο πιο σοβαρό ζήτημα πριν από μία ώρα περίπου όταν μιλήσαμε για τις προβλέψεις δαπανών ε, και εσόδων πολλοί μίλησαν για την ε, κυβερνοασφάλεια και το ανοιχτό ασύρματο δίκτυο είναι ζήτημα κυβερνοασφάλειας. Πηγαίνετε σε ένα δωρεάν ε, Wi-Fi Καμιά φορά υπάρχει μία μέθοδος ε, που πρέπει να κάνει κανείς εγγραφή με το facebook ε, το όνομά του και το συνθηματικό του και αν ε, είναι σπασμένο τότε όλες οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται από εκεί ότι έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα όταν μιλάμε για ε, ελεύθερο Wi-Fi. Και είναι ασφαλές ε, δωρεάν Wi-Fi, που είναι μια καλή ιδέα νομίζω. Τότε ε, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πόσα και τάξεις μεγεθών μια φορά βοηθάει λίγο να σκεφτόμαστε το, το τι σημαίνουν αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα. Θα... δώσει κάποια στοιχεία στην Επιτροπή. Κύριε Χρυστοφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμεί θεωρούμε ότι το δικαίωμα πρόσβαση στο ίντερνετ και το είπαμε πάρα πολλέ φορές είναι το δικαίωμα για όλους τους πολίτες και δεν έχουμε παρά να χαιρετήσουμε προτάσεις που βρίσκονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, έστω ως πρώτο βήμα, είναι προς την ορθή κατεύθυνση, γιατί θα επιτρέψει σε πολίτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμω πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά σε αυτόν τον τομέα να διαπρέψει. Δεν εννοείται ψηφιακή Ευρώπη, ενιαία ψηφιακή αγορά, χωρί να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα απομακρυσμένε χώρε και η δικιά μου χώρα είναι οι πιο απομακρυσμένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και νησιώτικοι και ιδιαίτερα οι νησιώτικε περιοχέ πραγματικά υποφέρουν από ανεπάρκεια σύνδεση με το WiFi αλλά και με ψηλό κόστο με χαμηλέ ταχύτητε. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και να δώσουμε αυτή την ισότιμη δυνατότητα σε όλου του πολίτε. Θεωρώ ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτά τα προγράμματα, αυτό το ευρώ πολλαπλασιάζεται ω επένδυση και επιστρέφει πίσω. Μειώνει τη γραφειοκρατία, αυξάνει τι θέσει εργασία, δημιουργεί πρόσβαση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ουσιαστικά δημιουργεί μια κοσμογονία. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να το βλέπει ω δαπάνη και έξοδο και θεωρώ ότι τα 120 εκατομμύρια που δίνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρία χρόνια είναι ανεπαρκέ. Λείπει εκείνο το όραμα που θα ανταποκρίνεται προ όλου και προ όλε τι χώρε. Ιδιαίτερα, όπω είπα, σε νησιώτικε απομακρυσμένε περιοχέ που θα μπορούσε εκεί να εφαρμοστεί πιλωτικά και να δοθεί δωρεάν Wi-Fi σε όλου και να αποδειχθεί για πρώτη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρο. Άκουγα τον ιδρυτή του Facebook να λέει ότι ο ίδιο προσωπικά θα παράσχει πρόσβαση σε όλου του Αμερικανού πολίτε οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο WiFi. Εάν ένα άνθρωπο μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι εδώ είναι μια σημαντική πρόκληση. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Στηρίζουμε το WiFi fi for EU και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φανεί πιο γενναιόδορη προ αυτή την κατεύθυνση. Όπω τόνισα, δεν είναι δαπάνη. Δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση και οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία που έχει και οικονομικό χαρακτήρα και επενδυτικό και κοινωνικό και το πιο σημαντικό συνδέει πλέον ολόκληρη την Ευρώπη και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και μέσα στα πλαίσια και της γενικότερης πολιτικής που ανέπτυξε πολύ ορθά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Γιούγκερ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ασχολείται με τα ασήμαντα, πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί με τα σημαντικά. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο στρατηγικής σημασίας και τα 120 εκατομμύρια θεωρώ ότι σε τρία χρόνια θα αρθούμε το 2019 και θα παραδεχτούμε όλοι ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Άρα θεωρώ από τώρα πρέπει να αναθεωρήσει τον οικονομικό στόχο, να τον επαυξήσει, να τον πολλαπλασιάσει και είμαι βέβαιος ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ κάτι αλλάζει και είμαστε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μπορεί να θεωρούν οι πολίτες. Monsieur Negrescu. Thank you και εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία και βεβαίως ο συνάδελφος είπε ότι ε, δίνουμε λίγα λεφτά που δεν αρκούν για αυτό το σημαντικό έργο. Να προσθέσω κάποια πράγματα. Τέσσερα. Πρώτα απ' όλα πρέπει όντως να βελτιωθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές αλλά να βελτιωθούν και οι συνδέσεις ε, σε περιοχές όπου ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ε, διαδίκτυο. Πρέπει δηλαδή να ληφθεί υπόψη και η κοινωνική ανισότητα, όχι μόνο η γεωγραφική ε, διάσταση. Δεύτερον, να φροντίσουμε να μην επενδύουμε σε Συνδέσει ασύρματο διαδικτύου εκεί που είχαμε ήδη επενδύσει σε κάτι τέτοιο. Γιατί είχαμε ήδη επενδύσει σε διάφορε πόλει για δωρεάν ε, διαδίκτυο και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την πρόσβαση σε δίκτυο σε άλλε κοινότητε. Τρίτον, θεωρώ ότι μαζί με αυτό το έργο πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη ψηφιακή εκπαίδευση. Ένα συνάδελφο ανέφερε την ανάγκη κυβερνοασφάλεια. Ε, δεν ανάγκη τόσο μακριά. Εργαζόμουν στον κλάδο, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε αλλά η ψηφιακή εκπαίδευση βεβαίως θα πρέπει να περιλάβει την συνδεσιμότητα και τέταρτον το θέμα της εφορίας. Δημιουργούμε μια σύνδεση, μπορεί να είναι καλό δίκτυο για ένα, δύο, τρία χρόνια, αλλά μετά τι γίνεται. Πρέπει να το αντικαταστήσουμε, ποιος θα το αντικαταστήσει ή να το κλείσουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα της βιωσιμότητας, γιατί Δυστυχώ, αν δεν επενδύσουμε αρκετά, θα απαξιωθούν αυτά τα λεφτά σε λίγο καιρό. Ευχαριστώ, κύριε Ζούμπιχ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σημαντική έκθεση. Πρέπει νομίζω να προσέξουμε να υπάρχει εδώ πέρα τεχνολογική ουδετερότητα. Έχουμε αφενός ε, το θέμα της ε, πέμπτης ε, γενιάς ε, των τηλεπικοινωνιών ε, που θα αναπτυχθεί και από την άλλη βεβαίως έχουμε το θέμα του ασύρματου δικτύου. Οπότε έχουμε τις τηλεπικοινωνίες που έχουν πολύ ισχυρή ρύθμιση ενώ το ασύρματο διαδίκτυο δεν έχει τόση έπιση. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να διατεθούν προφανώς με δημόσιο διαγωνισμό, με διαφάνεια και θα πρέπει να πάνε και σε μικρές ε, και μεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα μικρές επιχειρήσεις να κάνουν ε, επιτόπια τις εγκαταστάσεις και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Τόρβαλτς γιατί βεβαίως οι πολίτες πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις εκεί πέρα ε, και θα συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα και δεν θα υπάρχει hacking σε αυτές τις συνδέσεις. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη στην προκήρυξη των, διαγωνισμών, να είναι υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σκέφτηκα στην προηγούμενη συζήτηση όταν κοιτάζαμε τα πιλωτικά έργα ότι όταν μιλάμε για χρηματοδότηση πρέπει να κοιτάμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, εάν κάτι είναι κατάλληλη χρήση των χρημάτων ε, των φορολογουμένων. Δεύτερον, ε, υπάρχει πραγματικός λόγος που δεν γίνεται κάτι σε επίπεδο κράτους μέλους. Τρίτον, εάν θα έχει πραγματική αξία σε σχέση με τη δαπάνη. Και υπήρχαν ε, κάποια έργα για τα οποία δεν θεωρούσα ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, όταν μιλάμε για δημόσια σύρματα δίκτυα, Νομίζω ότι εντάξει, κάτι μπορούμε να πούμε, ότι μπορεί να γίνει κάτι με χρήματα των φορολογουμένων, αλλά δεν βλέπω την ανάγκη να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τα κράτη-μέλη. Να παρέχουν τα κράτη-μέλη δωρεάν Wi-Fi αν θεωρούν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Έχω επίση μια ανησυχία όσον αφορά την ανάγκη για τέτοια έργα. Δηλαδή προσωπικά εγώ χρησιμοποιώντας ε, το Wi-Fi πριν από λίγα χρόνια το Wi-Fi σε δημόσιους χώρους ε, θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια όταν έχετε κάποιος με το κινητό του και δεν έχει δεδομένα στο κινητό. Σήμερα όμως θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα θα έχουν δεδομένα στο κινητό τους και αναρωτιέμαι πραγματικά εάν είναι σωστή η χρήση χρημάτων αυτή σήμερα σε σχέση με, πέντε, με πριν από 5 ή 10 χρόνια. Και τέλος μιλάμε εδώ για ένα κονδύλι πέρα από τον έξτρα δηλαδή που θα προσθεθεί στον κοινωτικό προπολογισμό και αυτό νομίζω είναι μια ανησυχία. Σας ευχαριστώ. Ο Ράιμερ Μπέγκε και πάλι τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση που πρέπει να γίνει και βεβαίως σχετίζεται με τη συζήτηση για έτσι, κάπως ε, ισότιμες ε, συνθήκες ζωής και ευκαιρίες ε, μεταξύ των πόλεων και των απομακρυσμένων περιφερειών. Επίσης πρέπει να γίνει μια διάκριση η συζήτηση του τι σημαίνει διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους. Καλό είναι να γίνει αυτό. Και Βεβαίω, ε, εκτός Ευρώπης ε, έβλεπε κανείς ότι σε κάποια ξενοδοχεία ήταν καλύτερη σύνδεση από ότι ε, σε περιοχές της χώρας μου. Και τώρα βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να απολυθούν σπίτια γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και πλέον εννοούμε και την σύνδεση στις υποδομές και ποιο ήταν... Ε, έχουμε παραδείγματο χάρη ε, ένα παράδειγμα ενός χωριού 700 ατόμων ε, λίγα χιλιόμετρα βορείως του Αμβούργου για το οποίο δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τις λεπικοινωνιακές εταιρείες και περιμένουν χρόνια για να αποκτήσουν μια γρήγορη σύνθεση. Δεν έχει νόημα τώρα βεβαίω να λέμε για διαρθρωτικά τα κτλ. Μιλάμε για τελείως διαφορετική διάσταση του θέματος. Μιλάμε για την ε, περίπτωση αυτή που σας λέω τα χωριά αυτά μαζεύτηκαν μερικά χωριά μεταξύ 700 και 2.000 κατοίκων και τελικά έκαναν μεταξύ τους έναν συνεταιρισμό και χρηματοδότησαν μία σύνδεση η οποία βεβαίως ε, τους συνέδεσε με τον έξω κόσμο και βεβαίως ε, υπάρχει και το θέμα και των ε, οπτικών ινών και βεβαίως αυξήθηκε θα έλεγα γενικά και η ποιότητα ζωής τους. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία στις δομές, στις περιοχές αυτές να διαφυλάξουμε και ίσως και να κερδίσουμε κάτι περισσότερο. Αλλά αυτό σημαίνει και δική μας πρωτοβουλία και συνεργασία με ενώσεις ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις με βάση σωστές προτεραιότητες. Και βεβαίως μπορούμε να δώσουμε κάποια κονδύλια που μπορούν να υποστηρίξουν, αλλά ας μην περιμένουμε για να ξεκινήσει αυτή η δουλειά τον ευρωπαϊκό Περιφερειακό Προϋπολογισμό να διαθέσει τα κονδύλια. Πρέπει να γίνει ή κάποιον εθνικό ή τοπικό προυπολογισμο περιφερειακό προυπολογισμο να διαθέσει τα κονδύλια. Πρέπει να γίνει δουλειά. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Ο κύριος Σίκοφτς και τελευταίος. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Μια και σύντομα θα περάσουμε στη ψηφοφορία, θα είμαι σύντομος. Είμαι κυνηγό, μου αρέσει να περπατάω στο δάσος και πολλές φορές βλέπω ότι στα δάση η κάλυψη του, της σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι πολύ γρήγορη και πολύ καλή θα έπρεπε να υπάρχει το διαδίκτυο, μάλλον εκεί που ζει ο άνθρωπος όμως και όχι εκεί όπου ζουν τα ζώα, γιατί δεν γνωρίζω κανένα αγριογούρουν όπου να υποφελείται του υπερταχέως διαδικτύου. Σε ορισμένε περιοχέ, λοιπόν, έχουν δοθεί και επιδοτήσει από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για τη βελτίωση τη συνδεσιμότητα στην Ήπεθρο. Και εγώ θα έλεγα ότι προσωπικώς το γρήγορο διαδίκτυο στο δάσος δεν το χρειάζομαι. Θα παρακαλέσω λοιπόν την Επιτροπή τις αρχές της ε, καλής διασύνδεσης και συνδεσιμότητας να τις ε, επικεντρώσει στις πόλεις και όχι στα δάση όπου μάλλον τα ζώα μας ενδιαφέρει να απολαμβάνουμε παρά το διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος, ναι, ίσως όμως με το μένα ένα καλό διαδίκτυο να προειδοποιούνται τα ζώα ότι φτάνουν κυνηγοί για να φύγουν τρέχοντας. Εν πάση περιπτώσει, καλή επένδυση. Μπορεί και τα ταμεία συνοχής να συμβάλλουν για τον σχετικό εξοπλισμό. Άπαξ βέβαια και προσδιορίσουν τη σχετική προτεραιότητα οι τοπικές αρχές. Και ασφαλώς η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει προς ε, και μαζικές επενδύσεις και για το διάστημα και για τους δορυφόρους, για πυκνότερη δορυφορική διασύνδεση. Κυρία Μυριάντα, παρακαλώ πολύ σύντομα για να ολοκληρώσουμε. Ναι, πολύ σύντομα και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος από οποιαδήποτε κυβερνοαπειλή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, το παρακολουθούν και να επιβλέπουν οι τοπικές αρχές. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία δηλαδή να μην το υποστηρίξουμε. Επίσης πρέπει, συμφωνώ, να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας στις πιο υποβαθμισμένες και φτωχές περιοχές, ε, πακέτα με όγκους δεδομένων που δεν χρειάζεται κανείς, αναφέρθηκε νωρίτερα. Ναι, αλλά κοιτάξτε λίγο, κάποιοι δεν έχουν ούτε αρκετά για να βάλουν φαγητό στο πιάτο ή να βάλουν πετρέλαιο στο λέβητα. Ε, τι να το κάνουν λοιπόν το πακέτο με φτηνό όγκο δεδομένων ή δωρεάν όγκο δεδομένων. Για να τους βοηθήσουμε να ξεφύγουν από την παγίδα της ε, φτώχειας πρέπει να κάνουμε μια επένδυση που δεν είναι μεγάλη, δεν είναι τεράστιο έξοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τεράστια σημασία σε επένδυση. Ε, σημειώνω λοιπόν όλε τι παρατηρήσει και το σχόλιο τελευταίου συναδέλφου για το δάσο. Να σα πω κάτι. Αν τυχόν ε, σα τύχει και παραβατήσετε και σπάσετε το πόδι σα ή έχετε κάποιο άλλο ατύχημα, χρειάζεστε καλή πρόσβαση. Εν πάση περιπτώσει, α αφήσουμε τα αστεία. Το θέμα δεν είναι να συνδεθούν οι απομακρυσμένε περιοχέ, οι δασικέ τη υπαίθρου, αλλά οι μικρέ ε, οι μικροί και απομακρυσμένοι οικισμοί στην Ήπεθρο που δεν έχουν καλή διασύνδεση. Αυτό ήταν ο στόχο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με το σχόλιο όλων θα έχουν μια πολύ καλή έκθεση. Ε. Να χαθεί το δάσο φυσικά. Λοιπόν, όσοι θέλουν να καταθέσουν τροπολογίε την 9η Μαρτίου 12η μεσημβρινή η προθεσμία. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει την 3η Απριλίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή επί την Επιτροπή Ήτρε δηλαδή, στις 25 Απριλίου. Συνάδελφοι, θα περάσουμε τώρα σε ψηφοφορίες. Σας ζητώ να χρησιμοποιήσετε όλοι τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να κάνουμε μια δοκιμή καταρχάς. Άρχεται η ψηφοφορία. σε κάποιους δεν λειτουργεί. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση πρακτική. Όταν βλέπω εδώ τον κατάλογο των ψηφοφοριών, θα ήθελα να μου πείτε αν τις εβδομάδες που προηγήθηκαν είχατε κάνει ένα διαγωνισμό ποιος θα καταθέσει τις περισσότερες τροπολογίες Υπάρχει μία συνάδελφος που παρουσίασε 501 τροπολογίες. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν να υπήρχε ένας διαγωνισμός. Τώρα γιατί μας τις δώσατε αυτές τις τροπολογίες, θα τις ψηφίσουμε. Λοιπόν, ε, τέλος της ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δοκιμής. Ίσως ε, θα υπάρξει δυνατότητα να ψηφίσουμε ο μπλοκ ομαδών εφόσον θέλετε να κερδίσουμε κάποιο χρόνο εφόσον ε, οι τροπολογίες έχουν τον ίδιο στόχο, σαν παράδειγμα την διαγραφή κάποιων τμήματων ε, του ε, κειμένου. Και για τα άρθρα όπως και για την αιτιολογική σκέψη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα για την έκθεση του κυρίου Άσχουαρθ για την προετοιμασία του προπολογισμού τρίτο τμήμα. Υπάρχει καταρχάς το 1α συμβιβαστική πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Compromis 1B. Qui est favorable. 1β. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 43. Ποιοι είναι υπέρ. 43 d'abord, si vous voulez bien. 43 παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 54 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία τώρα. για έρευνα, υποδομές για τις μικρομεσαίες κτλ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 69. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ογδόντα πέντε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 92 λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 ποιοι είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 108 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές και θα δώσω τώρα τον λόγο ε, στον εισηγητή για την 8. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την συμβιβαστική 8 υπάρχει μία μικρή προφορική τροπολογία. Πρέπει να βάλουμε την λέξη στα αγγλικά especially ανάμεσα στο υψηλές κοινωνικές επιπτώσεις και στις περιφέρειες. Θα πρέπει να βάλουμε βασικά την λέξη especially. Το υπόλοιπο μένει ως έχει. Λοιπόν, για την συμβιβαστική 8, μαζί με την προφορική τροπολόγηση την οποία έκανε ο εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10. Όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 134. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 139 σε τέσσερα τμήματα. αλλά έχει γίνει δεκτή εν συμβιβαστική 10, οπότε το πρώτο τμήμα καταπίπτει, παραμένει το δεύτερο τμήμα, που είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τρίτο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τέταρτο τμήμα έχει και αυτό καταπέσει. 149 υπέρ κατά δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για το 149 άρχεται η ψηφοφορία πέρα στις ψηφοφορίες απερίφθη 19 κατά 13 υπέρ 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 13 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 184 υπέρ κατά αποχές δεκτή 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 228 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 230 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 232 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 2.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.38 υπέρ κατά αποχές 2.39 υπέρ κατά για το 2.38 ξανακάνουμε την ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 2.41 ποιοι είναι υπέρ Διακόπτει ο πρόεδρος. 2.39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.41. 2.40 μάλλον. Διορθώνει ξανά ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.44 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.44. Α, όχι. Ψηφίστηκε το 2.44. 2.45 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 267 έχει αποσυρθεί 268 υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2,70 υπέρ. Συγγνώμη, 2,69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 2.72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σας προτείνω 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 να ψηφιστούν ομαδικά παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τώρα επί του συνόλου του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές, συγχαρητήρια στον Γενικό Εισηγητή. Θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Πόνς για τη διαχείριση των αλλιευτικών στόλων στις απότερες περιφερειακές ζώνες. Καταρχάς για την τροπολογία 4 και την τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι δύο τροπολογίες αυτές απορρίπτονται. Οι έξι υπέρ κατά αποχές δεκτές. Επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 8 ψηφίζεται Πέραστη ψηφοφορίας απορρίπτεται 19 υπέρ 12 κατά 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Επί του συνόλου του κειμένου τώρα, ονομαστική κλίση. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 3 ε, κατά μία αποχή συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα ερχόμαστε στην έκθεση Ντεπρέ. αναβάλλεται η ψηφοφορία σας για το μήνα Απρίλιο. Το είχα πει άλλωστε στην αρχή της συνεδρίασης. Έχουμε 501 τροπολογίες για την έκθεση Gerard Depré, λέει ο πρόεδρος, σχετικά με το Eurodac. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω, μιας και έχουμε ορισμένες τροπολογίες της κυρίας Μοντέλ, οι οποίες είναι, έχουν σαν στόχο αποκλειστικά τη διαγραφή και σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό νομίζω ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια ενιαία ψήφος επί του συνόλου των τροπολογιών Μοντέλ. Η πρότασή μου μπορεί να γίνει δεκτή. Είναι κάποιος κατά της ενιαίας ψήφου, ποιοι είναι υπέρ της προτάσεως αυτής, ποιοι είναι κατά, συνεπώς. κύριε Άρνοτ, έχετε ζητήσει το λόγο. Διερωτώ γιατί να κατεθούν 500 ε, τροπολογίες και να μην ψηφίσετε τελικά το κείμενο. Τόση φασαρία για το τίποτα δηλαδή. Ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε. Όμου, το σύνολο των άρθρων, το κατάλογο τον έχετε. Και αρχίζουμε με την 84. Για να τελειώσουμε στη σελίδα 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθησαν. Τα ίδια προτείνω για την ψηφοφορία στις αιτιολογικές σκέψεις. Σελίδα 25-26. Μέχρι τα μισά της 26. Ξεκινούμε με την τροπολογία υπαριθμών 17 και τελειώνουμε με την 83. Την ψηφοφορία μπλοκ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές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 κατά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 19 υπέρ 13 κατά 13 υπέρ κατά Να σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ. Η 13 τώρα. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 13 κατά. Ετυλογικές σκέψεις, τροπολογία 14 υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη. 15 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 16 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 19 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. Υπαριθμόν 1 υπέρ, κατά. απερίφθη 21 υπέρ, κατά. Απερίφθη 2 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά δεν βλέπω να σηκώνει τα χέρια σας όλοι επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 26 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 13 κατά. Ήταν 26 αυτή. Υπαριθμών 5 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 31 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε τη 31 ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας. Και εγκρίνεται 17 υπέρ, 14 κατά. 35 υπέρ, κατά. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 20 ψήφι κατά, 12 υπέρ. Να σηκώνω το μασκρά το χέρι. Τροπολογία 6 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται... Αλλά στο επαληθεύσουμε... Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 18 υπέρ, 14 κατά. Το σύνολο της προτάσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ. 13 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα έχουμε να ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Καρθίας Σαββόλ Ταμείο Συνοχής, εξορρόπηση μεταξύ των χρηματοοικονομικών μέσων και των πιστώσεων. Συμβαστική παριθμόνα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, απερίφθη. Δέκα, υπέρ, κατά. Μάλλον έχει απερίφθει. Ας επαληθεύσουμε όμως, δέκα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 16 κατά, μία ψήφος, 15 ε, υπέρ. Και αυτά είναι οι 10. 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 21 υπέρ, κατά, αποχές. Απερίφθη. 4. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ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 και εγκρίνεται 28 υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Και συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Τρίτο τμήμα του προπολογισμού. Δεν έχουμε αιτήματα για εμβάσματα. Στα άλλα τμήματα του 17 έχουμε τον κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουμε να πληρώσουμε αποζημίωση προς μια εταιρεία που κέρδισε δίκη εις βάρος επιτροπής. Ευτυχώς μπορέσαμε τα χρήματα αυτά να τα αντλήσουμε από αμοιβέ και αποζημιώσεις και παρακαλώ την Επιτροπή να εγκρίνει ή να σας εξηγήσω πρώτα τι ζητάει η Ombudsman που είναι ένα άλλο θέμα. Όχι, στο πρώτο θέμα. Θέλει κανείς ε, να ρωτήσει κάτι στον συγκητή μας ή να αμφισβητήσει. Όχι. Από ό,τι βλέπω. Πρώτο αίτημα λοιπόν για έμβασμα. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Όχι. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Όχι, γιατί δεν χρειάζεται ψηφοφορία. Είναι μικρά τα ποσά, στο εγκρίνουμε. Δεύτερο έμβασμα, κύριε Τάραντ. Ευελτιώνει το η δεύτερη αυτή πρόταση την ευελιξία στο γραφείο της Ομπλουσμαν και είναι και πολύ μικρό το ποσό. Μια μόνιμη θέση απασχόληση μετατρέπεται σε προσωρινή. Δεν θα κάνει εξηγήσει. Όχι. Τότε δεν χρειάζεται ψηφοφορία εφόσον δεν εκφράζει κανείς αντίρρηση. Η κυρία Χολμάιερ θα μπορούσε να μας παρουσιάσει ίσως ε, μία έκθεση για τη Frontex και το κτηριακό, αλλά δεν έχει ακόμα τα στοιχεία νομίζω στη διάθεσή της ώστε να καταλήξει στη διατύπωση γνωμοδότης, άρα η ψηφοφορία αναβάλλεται και έτσι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας και επισημαίνω κάποιες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την προσεχή μας τακτική συνεδρίαση στις 20 και 21 Μαρτίου που θα ακολουθήσει μία ακόμη στις 27 στις 6 και 30 και αντίστοιχα ματαιώνεται η συνεδρίαση της 30 Μαρτίου. Σημειώστε αυτές τις αλλαγές παρακαλώ στην, στην ατζέντα σας. Δεν βλέπω να είστε κανείς άλλο στο λόγο και αν δεν έχετε κι εσείς καμία ερώτηση ή παρατήρηση μπορώ να κηρύξω το πέρας της συνεδρίασης ευχαριστώντας σας για την πολύ καλή συμμετοχή και επόμενος καλό βράδυ.